Ε, good morning everybody. Καλή σας μέρα. Αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Πρόκειται για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η σύμβαση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ε, κατακολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών. Έχουμε ήδη κάνει δύο δημόσιες ακροάσεις στην Επιτροπή μας και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ειδικού εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό, καθώς επίσης και την άποψη των ε, θεσμικών παραγόντων. Σήμερα θα ακούσουμε πάλι τα βασικά στοιχεία της σχετικής έκθεσης και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Νταλόν Μπονεφουά Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με περηφάνεια σήμερα σας παρουσιάζω την έκθεση πρωτοβουλία μας, την προσωρινή έκθεση πρωτοβουλία μας για την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοικογενειακής βίας. Πρόκειται για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Κάποια στοιχεία για τη Σύμβαση αυτή που εγκρίθηκε στις 7 Απριλίου του 2011. Είναι το πρώτο διεθνές μέσο δεσμευτικό νομικά για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών η σεξουαλική παρενόχληση, η βία, η σωματική και ψυχολογική βία, όλα αυτά αποτελούν πράξεις βίας. Και συνήθως οι θύτες είναι οι άντρες και τα περισσότερα θύματα είναι οι γυναίκες. Πρόκειται δηλαδή για μια βία η οποία είναι συνάρτηση του φίλου και απορρέει από την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάτι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που σπάνια καταγγέλλεται. Έτσι λοιπόν χρειαζόταν ένα νομικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια, να υπάρχει μια πολυδιάστατη προσέγγιση των τριών ΟΠΕ που είναι η πρόληψη, η προστασία και η δίωξη, που στα γαλλικά αρχίζει με ΠΕ βέβαια. Πρόκειται λοιπόν για την ευαισθητοποίηση, για την προστασία και την βοήθεια προς τα θύματα, όπως επίσης και τη δίωξη των θητών πρέπει να καταδικάσουμε όλες τις μορφές βίας σε βάρος των γυναικών. Και επιμένω σε κάτι σημαντικό, ότι στις νομικές ε, διαδικασίες μετά από τέτοιου είδους βία Συνήθως ε, λέμε ότι οι παραδόσεις ή η θρησκεία δικαιολογούν κάποιες τέτοιες πράξεις. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει ποτέ, γιατί ανεχόμαστε τη βία εξαιτία τέτοιων παραδόσεων θρησκευτικών ή άλλων. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν την αποτελεσματική εφαρμογή των όσων αναφέρει η Σύμβαση, προβλέπονται και ιδιαίτεροι μηχανισμοί. Όλα τα μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, αλλά μόνο 14 κράτη-μέλη έχουν κυρώσει κιόλα τη Σύμβαση αυτή. 14 Μαου του 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη σύμβαση αυτή. Θα υπάρξει έτσι ένα ε, συνεκτικό πλαίσιο νομικό για να προστατευτούν οι γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κύρωση εκ παραλίλου και από όλε τι χώρε μέλη. Πηγαίνετε στη σελίδα 7 τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητε. Η πρόταση αυτή συζητιέται στο Συμβούλιο επί του παρόντος και όταν υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και εκείνο να εγκρίνει το κείμενο. Προηγουμένως όμως πρέπει να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή πρωτοβουλίας για να δηλώσουμε ποιε είναι οι δικές μας οι προτερότητε. Το έργο μας με την Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλ που είναι η συγγήτρια από πλευράς της Επιτροπής Γυναικών είναι πολύ απαιτητικό και θέλω να επιμείνω σε κάποια σημεία της έκθεσης αυτής. Πρώτον, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών πρέπει να είναι ευρύτερη δυνατόν και χωρίς επιφυλάξεις. Δεν αποκλείονται οι χώρες μέλη από τις δικές τους αρμοδιότητες μεμονωμένα. 14 μόνο έχουν κυρώσει και δεν φτάνει. Έπειτα, η συνολική προσέγγιση, πολύ διάστατη τη σύμβαση αυτή, είναι επίση κάτι αναγκαίο για να απαλληθεί πλήρω η βία σε βάρο των γυναικών. Επιμένουμε στην αλλαγή νοοτροπία από πλευρά ολόκληρη τη κοινωνία. Ω εισηγήτρια εκ μέρου τη ΛΥΜΠΕ, λοιπόν, δίνω μεγάλη σημασία στι διατάξει που αναφέρονται για την μετανάστευση και υπενθυμίζουμε ότι οι μετανάστε και τούντε άσυλο είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη βία που απορρέει από το φύλλο και είναι μια βία η οποία εκλαμβάνεται ως δίωξη σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενέβης του 1951. Ζητούμε από τις χώρες μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη το φύλλο κάθε φορά που εξετάζουν μια αίτηση ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται και να συμμετέχει είτε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο, είτε κατά τη διάρκεια του μηχανισμού παρακολούθησης. Και άπαξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει προσχωρήσει στην σύμβαση. Η εφαρμογή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξουν κατάλληλοι πόροι για να πετύχει η εφαρμογή. Ζητάμε από την Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη. Μία οδηγία, για παράδειγμα, η οποία θα περιλαμβάνει κοινού ορισμού για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη βία σε βάρο των γυναικών και θα βοηθήσει να ενισχυθεί το αποτέλεσμα τη σύμβαση αυτή. Η προσχώρησή μα είναι ένα πρώτο βήμα. Η μάχη μα δεν σταματάει με αυτήν την προσωρινή έκθεση. Η προσχώρηση τη Ένωση είναι ένα ισχυρό πολιτικό βήμα που δηλώνει την επιθυμία Τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάλληψη τη βίας σε βάρο των γυναικών. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κορέτσα Μπίλτ και στους σκιώδει εισηγητές. Θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση μας του Απριλίου, στι 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κορέτσα Μπίλτ, τη συνεισηγήτρια. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κριστίν, ε, Πραγματικά βρήκα πολύ ευχάριστη όλη την προπαρασκευαστική εργασία που κάναμε μαζί. Οργανώσαμε και μια σειρά ακροάσεων το Νοέμβριο, το Μάρτιο και στις δύο επιτροπές και το Policy Department μας βοήθησε πάρα πολύ με το εργαστήριο που αφορούσε την σημασία της συλλογή δεδομένων. Έτσι λοιπόν σήμερα παρουσιάζουμε μια μακρά και σβάθος δουλειά που κάναμε από κοινού. Όπως ε, είπε και η Κριστίν, η βία είναι ε, ευρέως ε, εξαπλωμένη στην Ευρώπη, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, είτε στο σπίτι, είτε δημοσίως, είτε στο διαδίκτυο. Οι γυναίκες διώκονται, παρενοχλούνται, βιάζονται, ξυλοκοπούνται. Δεν υπάρχει καμία κουλτούρα, καμία παράδοση, καμία θρησκεία που να δικαιολογεί τη βία η βία κατά των γυναικών ε, συχνά είναι βία ανδρών κατά των γυναικών και είναι σοβαρό έγκλημα. Και έτσι θα πρέπει να το μεταχειριστούμε. Γιατί κάνουμε όλο αυτό το έργο, όλη αυτή τη δουλειά. Γιατί η Σύμβαση της Κασταντινούπολης, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι το μόνο διεθνές μέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, που μας δίνει τα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε ε, τη βία και να προστατεύσουμε τα θύματα και να κάνουμε μακροπρόθεσμη δουλειά σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, να οικοδομήσουμε τις ικανότητες, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, να κρατήσουμε το θέμα στην ημερησία διάταξη και να αλλάξουμε την οτροπία και τον πολιτισμό. Στον κόσμο που ζούμε τώρα, από τον Πούτιν μέχρι τον Τραμπ, ο σεξισμός ε, πραγματικά κυριαρχεί και στο πολιτικό θεματολόγιο και υπάρχει μια σοβαρή παρεξήγηση για το ότι υπερασπίζουν κάποιες ε, θρησκείες, ε, κάποιες κουλτούρες, ότι παραδείγματο χάρη το σώμα των γυναικών ουσιαστικά αποτελεί τη μονάδα μέτρησης για την ηθική των ανθρώπων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε μια ευκαιρία ευκαιρία εδώ με την προσχώρηση στη σύμβαση να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα. Είπες και εσύ Κριστίν, πολύ πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν καν ακυρώσει τη συνθήκη και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν επικυρώσει θα εργαστούν προς ε, την κατεύθυνση αυτή, παρά να μας λένε ότι τα κράτη τους ε, δεν έχουν κυρώσει τις συνθήκες. Εμείς ε, δεν θα ακολουθήσουμε τις κυβερνήσεις μας, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις μας, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, όταν πρόκειται να υπερασπίσουμε τις γυναίκες θύματα βίας. Χτες ε, είδαμε ότι ε, πάνω από 70 εκατομμύρια κορίτσια σήμερα στην Ευρώπη ακόμη που ουσιαστικά δίνονται ε, σε άνδρες για να τους πεντρευτούν, σε άνδρες που δεν τους έχουν ξαναδεί ποτέ πριν. Τους κλέβουν την παιδική τους ηλικία. Μόνο στη Σουηδία έχουμε πάνω από 130 κορίτσια που ήδη τα έχουν παντρέψει. Ευχαριστώ την Κομισιόν που παρουσίασε την πρόταση αυτή και για τη δουλειά που κάνει και την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που κάνει πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την ε, ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και καλό τα κρατημέλη να συνεργαστούν περισσότερο μαζί του και με τη Eurostat. Χρειαζόμαστε πιο σαφή δεδομένα για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το θέμα στην μερσία διάταξη. Επίσης, θέλω να αναφερθώ στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι πολύ σημαντική και εκτιμώ τη συνεργασία που έχουμε σε ό,τι αφορά την, στην εφαρμογή της οδηγίας. Έχουν υπάρξει κάποιες ανησυχίες για το ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πολύ βραδείς ρυθμούς την οδηγία και θέλουμε λοιπόν να απευθύνουμε νέα έκκληση, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να επιδοθούν σε πιο επικοδομητικό και σβάθος διάλογο για τις επιφυλάξεις που έχουν ε, θέσει κάποια κρατημέλη. Ανάφερες Κριστίν κάποια επιφύλαξη για το άσυλο, αλλά και σε το θέμα του ορισμού του φύλου, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη υπερεξήγηση. Το φύλο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ζητήσαμε πολλές φορές, ε, σημαίνει τι ε, ουσιαστικά η βία, ε, η ενδοκογενειακή βία, η έμφυλη βία συμβαίνει κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες. Ε, βλέπουμε βία κατά των κοριτσιών, όχι κατά των αγοριών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε και την εφαρμογή όλων των υπόλοιπων νομοθετημάτων που έχουμε ήδη και θέλω να τα υπενθυμίσω εδώ, γιατί είναι αυτά μια ολιστική προσέγγιση για την καταπολέμηση τη βία στην οδηγία κατά τη εμπορία ανθρώπων, το Ευρωπαϊκή Διαταγή Προστασία, η οδηγία τη καταπολέμηση σεξουαλική κατοποίηση, η προστασία των θυμάτων, η οδηγία για την προστασία των θυμάτων. Σε όλα αυτά τα θέματα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σου, Κριστίν, και του υπόλοιπου Σκιώδη ε, και είμαι διαθέσιμη για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε. Και ίσω να προσθέσω κάτι ε, για λογαριασμό τη κυρία Ματέρα, η οποία είναι Σκιώδη ε, του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ τις δύο συνεισηγήτριες. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Να ξεκινήσουμε με τη σκιώδη του ΕΛΚ. Παρακαλώ, αν ε, θέλετε το λόγο, να κάνετε ένα λεύμα. Θέλεις ε, ξανά το λόγο, Μαρία. Ίσως να ξαναπάρω το λόγο αφού ακούσουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Η Χέλγα Στίβενς είναι σκιώδης από τη ΣΥΑΡ. Ίσως πρέπει να πάρει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω ε, τις ε, συνεισηγήτριες για το έργο τους ε, και την έκθεσή τους. Υποστηρίζω γενικά την πρωτοβουλία, όμως θα ήθελα τα σχολεία μου να είναι περιορισμένα και συγκεκριμένα. Η μεγαλύτερη μου ανησυχία ε, σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία είναι ότι δεν βλέπω καμία αναφορά στα άτομα με αναπηρίες παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες. Κατά τα άλλα όμως, ε, αναφέρεται ε, σε ένα σημείο, όμως κατά τα άλλα δεν υπάρχει αναφορά για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία και αυτό αποτελεί ντροπή. Επειδή λοιπόν ε, τα άτομα με αναπηρία, οι γυναίκες με αναπηρία κινδυνεύουν ιδιαίτερως ε, να βιώσουν ε, περισσότερη βία με μια μισή φορά παραπάνω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Στις, στην έκθεση, στην παράγραφο 5i, αναφέρονται οι ευάλωτοι άνθρωποι ε, και αποκλείονται και αναφέρονται μονάχα τα ε, παιδιά. Ε, όμως δεν γίνεται αναφορά στα παιδιά με αναφυρία και με ειδικές ανάγκες. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να τονίσω το άρθρο 4 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την μη διάκριση και την ισότητα, καθώς επίσης και την παράγραφο εδώ πέρα, η εφαρμογή ε, των πλαισίων της σύμβασης αυτής ε, από τα μέρη και συγκεκριμένα ε, μέτρα για την προστασία των θυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται χωρίς διάκριση, όπως είναι για παράδειγμα το φύλλο, το χρώμα, η θρησκεία, οι πολιτικές απόψεις, αλλά και ε, η εθνοτική καταγωγή. Και ε, ασχέτως ε, της καταγωγής, των σεξουαλικών προτιμήσεων, το επίπεδο υγείας, της αναπηρίας, το, ε, το καθεστώς μεταναστευτικό ή ασύλου και όπως βλέπετε λοιπόν η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη αναφορά στις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία και γι' αυτό το λόγο ε, ανυπομονώ να συνεργαστούμε με τις συγκήτριες ε, ούτως ώστε το, η πρόταση του Κοινοβουλίου ε, να, λαφ, να ληφθεί υπόψη και η σύμβαση να μπορεί να ε, εγκριθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Μίλνα. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες ήταν ε, μεγάλη ικανοποίηση να συνεργαστώ μαζί σας. Νομίζω ότι η Σύμβαση είναι ε, ένα εξαιρετικό νομοθέτημα. Επομένως, ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα να ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι εξαιρετική σύμβαση γιατί ορίζει ουσιαστικά την έμφυλη αλλά και τη βία κατά των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ. Και ουσιαστικά εδώ μιλάμε για μια σιωπηρή απειλή κατά των γυναικών, καθώς πρόκειται για σεξισμό. Είναι πάρα πολύ θετική η δουλειά που γίνεται για την υποστήριξη των θυμάτων και πρέπει ε, να γίνει δουλειά και σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό όποιος δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση αυτή να την κυρώσει πολύ σύντομα και να εκπονήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική, μια ευρωπαϊκή οδηγία για να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Έτσι λοιπόν, εγώ θα συνεργαστώ με τις συγγήτριες ε, για να καταθέσω κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εδώ εκπροσωπώ ε, την σκιώδη των Πρασίμων τόσο στη ΦΕΜ όσο και στη Λίβη και θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ε, για την συνεργασία και την, και την έκθεση και τις δύο συνεισηγήτριες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ε, σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και έχουμε πολλές κυβερνήσεις ε, ε, υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που δεν βλέπουν για ποιο λόγο θα πρέπει να έχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ευρία υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες να το θέσω έτσι. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε μια ισχυρή στάση απέναντι στη βία κατά των γυναικών ε, και ε, όσον αφορά την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή κράτη-μέλη όπως είναι για παράδειγμα η Πολωνία. Το Δεκέμβριο κάναμε μια καλή δήλωση για αυτό που ασκείται κριτική στην κυβέρνηση της Πολωνία, που λέει εντάξει ίσω θα το κάνουμε, ναι θα δούμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε εάν θα συμπεριληφθεί αυτό στην έκθεση ε, ώστε όσοι ε, έχουν επικυρώσει τη σύμβαση να την τηρήσουν κιόλα. Ε, και αυτό είναι το ιδιαίτερα σημαντικό. Ήταν κάτι που δεν είχαμε στο ε, παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και τα 14 κράτη-μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμα. Συμφωνώ με την Άννα Μαρία. Εμεί οι οποίοι καταγόμαστε από κράτη-μέλη και ιδιαίτερω εμεί που είμαστε κοντά στι κυβερνήσει αυτών των κρατών μελών που δεν τα έχουν επικυρώσει ακόμα, θα πρέπει να ε, πιέσουμε για να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, ε, θεωρώ ότι το Συμβούλιο ακόμα ε, μπλοκάρει ε, την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύμβαση και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το να πιέσουμε και ώστε να εγκριθεί, ότι, να αναγνωριστεί η βία κατά των γυναικών ως μια πολύ σημαντική παράβαση και ε, όσον αφορά την έκθεση της προηγούμενης ε, νομοθετικής περίοδου ήταν μια πολύ καλή ε, έκθεση αυτή τότε που απαιτούσε να υπάρξει μια νομοθετική πράξη κατά της ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη κατά της βίας κατά των γυναικών η Άννα Μαρία είπε ότι ο σεξισμός επίσης είναι ένας λόγος για τη βία κατά των γυναικών όμως θα πρέπει αυτό να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο στο κείμενο σε σχέση με το πώς είναι τώρα. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να συμπεριληφθεί είναι να ορίσουμε και να καταδικάσουμε τη βία κατά των γυναικών ως ένα πολύ σοβαρό έγκλημα και μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1993 είχαμε στη Βιέννη μια συνεδρίαση για τα, δικαιώματα των ε, για τα δικαιώματα των ανθρώπων και για πρώτη φορά αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό έγινε πριν από 20 περίπου χρόνια δηλαδή και πρόκειται λοιπόν μια από τις πιο σημαντικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Γενικά λοιπόν είναι μια πολύ καλή έκθεση και ευελπιστώ να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και να την περάσουμε και από την Ολομέλεια και να κάνουμε τόσο το Συμβουλίο όσο και τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η Μαρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ και συγχαίρω τις δύο συνεισηγήτριες για το ξέρω το έργο τους. Θέλω ευθύ αμέσω να πω ότι συμφωνώ. Όντω, έφτασε η ώρα οι χώρε μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψουν και να ακυρώσουν τη συμφωνία αυτή, τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και η έκθεση που εξετάζουμε σήμερα είναι πολύ σημαντική. Διέπεται από συνοχή, είναι ρεαλιστική και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα βήμα προς τα μπρος πραγματικά σε σχέση με τον τελικό μας στόχο που είναι η κύρωση της σύμβασης και η εκπόνηση και εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα προκοδοτούνται βέβαια από τους κατάλληλους πόρους. Θέλω όμως να επιμείνω σε ένα σημείο. Είναι σαφές ότι σήμερα κάποιες χώρες μέλη έχουν επιφυλάξεις για την ε, επικύρωση αυτή. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να έχουμε δράσεις που θα τις βοηθήσουν αυτές τις χώρες να ξεπεράσουν τους δισταγμούς τους. Ρεαλισμός είναι η λέξη κλειδί. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να σκεφτούμε για την εφαρμογή ενός συντονιστικού μηχανισμού που θα είναι αναγκαίος για την υλοποίηση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Κάποιες χώρες μέλη φοβούνται για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τη σύμβαση αυτή, γιατί όπως είπε και η Μαρία Κορέτσαμπίλ, πρόκειται για ένα μηχανισμό που είναι τελικό μόνος που διαθέτουμε και που θα επιτρέψει σε κάθε κρίκο της αλυσίδας να συνεισφέρει με θετικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει κάποιες χώρες. Γι' αυτό και επιμένω να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπως υπάρχουν σήμερα στις χώρες μέλη. Και μια ιδέα είναι ίσως να σκεφτούμε και την δημοσίευση κάποιων κατευθυντηρίων γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόληψη της βίας, με την στήριξη, την προστασία των θυμάτων, με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών αρχών, των δικαστικών αρχών που εξετάζουν τέτοιες υποθέσεις ή ακόμα να στηρίξουμε και την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων. Να λοιπόν, τέτοια συγκεκριμένα μέτρα είναι που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια να επιμείνουμε στις χώρες μέλη να ε, κυρώσουν και να μην έχουν πια δισταγμούς και φόβους που στο κάτω-κάτω είναι βάσιμοι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τις συνεισηγήτριες για το κείμενο που μας προτείνουν και ευχαριστώ και όλους τους συναδέρφους για την ένταση με την οποία θέλουν να μεταφέρουμε το μήνυμά μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ρέτσι Γκαρθία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ των Ευρωβουλευτών για την δέσμευση αυτή που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, βίας σε βάρος των γυναικών. Αναφέρθηκαν σημαντικά μέτρα που πιστεύω ότι όντω είναι αναγκαίο να εξεταστούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίγει η κύρωση από πλευράς του Συμβουλίου της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που εκπροσωπεί το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα οι χώρες μέλη που δεν έχουν ακόμα κυρώσει να το κάνουν. Αυτό όμω που είναι επίσης θεμελιώδες για να προχωρήσουμε στην πράξη αυτό που περισσότερο από μας θέλουμε, είναι να υπάρχει μια νομική βάση, ώστε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να νομοθετούμε. Αυτό είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για την ρήτρα γέφυρα, είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτή. Ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο έχουμε νομοθετική αρμοδιότητα, οπότε αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό βήμα προς τα μπρος. Αυτό θα κατοχύρωνε πρώτα απ' όλα την επιθυμία μας να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Οι γυναίκες στην Ευρώπη πρέπει να το καταλάβουν ότι δεν είναι μόνες τους, ότι στο πλευρό τους έχουν και τις χώρες μέλη, αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην καταπολέμηση ακριβώς της βίας σε βάρος τους. Μιλάμε για τρομοκρατία ματσιστική. Λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουν οι συμπεριφορές συνολικά, εγκάρσια, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην πρόληψη της βίας σε βάρος των γυναικών και αυτό να γίνει ήδη από τα σχολεία. Πρέπει λοιπόν όλοι όσοι έχουν κάποια αρμοδιότητα στο θέμα να μπορέσουν να δουλέψουν για να σταματήσει πια αυτή η τελευταία μάστιγα που έχουμε στην Ευρώπη και όχι μόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε συγχαρητήρια στις δύο εισηγητρίες για το έργο τους. Και ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους. Ό,τι προσπάθειες κάνουμε να καταλήξουμε σε κοινέ γραμμές για να πάψει πια αυτό το φαινόμενο της βίας σε βάρος των γυναικών είναι σημαντικά και μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το έργο μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κανέβα, παρακαλώ. Κυρία Κούνεβα, συγγνώμη, κυρία Κούνεβα. Χαίρομαι ιδιαίτερο που, αν και με καθυστέρηση, έχουμε στα χέρια μας το προσχέδιο έκθεσης για την σύναψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ευχαριστούμε τις ε, εισηγήτριες την κυρία Ρεβό και Κοράτσα για το πολύ καλό κείμενο που θα αποτελέσει η βάση για την δουλειά μας στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις προτάσεις και στις σκέψεις των συναδέλφων, από πλευρά μου υπάρχουν ορισμένοι τομείς που θα ήθελα να αναδείξουμε καλύτερα μέσα από το κείμενο της έκθεσης. Πρώτον, η πρόληψη, προστασία και υποστήριξη από κάθε μορφή βίας γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες όπως αναφέρει και η συνάδελφος. Προτείνω να υπάρχει ειδική μέρημνα για αυτήν την ευάλωτη κατηγορία πληθυσμού και βοήθεια να παρέχεται τόσο στις ίδιες όσο και για τις οικογένειές τους. Δεύτερον, πρέπει να ενδυναμώσουμε το κείμενο με προτάσεις για τη βία διαφόρων μορφών που ασκείται στο χώρο εργασίας. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιες την έχουμε βιώσει και ας δουλεύουμε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, η εφαρμογή χωρίς προγράμματα υποστήριξη και καμπάνιες ενημέρωσης δεν μπορεί να γίνει σωστά. Ζητάμε εκπαίδευση το προσωπικό που καλείται να διαχειριστεί θύματα βίας, γιατρούς, αστυνομικούς, ψυχολόγους και άλλοι κατηγορίες που τα εμπλέκουν, αλλά δεν ζητάμε κοντήλια για προγράμματα. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αναμασούν την καραμέλα του κόστους για την μία εφαρμογή της σύμβαση. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις που έχω, αλλά τα, περιοριστώ λόγω χρόνου. Εξάλλου θα τις κατατέσω με τη μορφή τροπολογιών. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι αισιόδοξη για την πορεία της έκθεσης για την εφαρμογή της σύμβασης. Και δεν σας κρύβω πώς περιμένω τη στιγμή που στην ερώτηση ποια είναι η πιο διαδεδομένα έγκλημα στον κόσμο, η απάντηση να μην είναι η βία κατά των γενικών. Εύχομαι καλή συνεργασία σε όλους και το καλύτερο αποτέλεσμα να βγάλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπεσέρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εκ μέρους ε, και τη Επιτροπή Γυναικών και εκ μέρου τη ΛΥΜΠΕ μιλάω, εκ μέρου τη ομάδα μου τη Άλντε. Και θέλω να ευχαριστήσω για το έργο του και την Αναμαρία και την Κριστίν. Και για το περιεχόμενο, αλλά και για την μορφή. Πραγματικά είναι θαυμαστό το έργο του. Δεν θέλω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θέλω όμω να πω μια σκέψη για την προέλευση και την αιτία η οποία μας οδήγησε στην έκθεση αυτή. Άρχισε να ισχύει πριν από τρία χρόνια η σύμβαση αυτή. Και πρέπει να αναγνωρίσω ότι από τη μια είμαι πολύ περήφανη που η πρώτη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν άρχισε η θητή αυτή ήταν ακριβώς να επιστήσει την προσοχή μας στην σύμβαση αυτή στη... για την οποία δεν είχε ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η αντίδραση της Επιτροπής Γυναικών ήταν πραγματικά όλοι ενωμένοι να στηρίξουμε την υπόθεση αυτή προκειμένου κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Και ακριβώ εδώ βρισκόμαστε, δυόμιση-τρία χρόνια σχεδόν μετά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενημερωμένη. Η κυρία Γιούροβε είπε ότι υπάρχει η βάση και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, κύρωση αυτή. Τώρα, εδώ και ένα χρόνο όμως περιμένουμε να προχωρήσει το Συμβούλιο. Είπα ότι είμαι περήφανη από τη μια και είμαι περήφανη γιατί και η ομάδα μου άλλη έκανε πολλά για να προχωρήσει η υπόθεση. Από την άλλη μεριά είμαι και απογοητευμένη γιατί πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό, τόσο δίκαιο, τόσο καλό, τόσο ολκυστικό στο κάτω-κάτω που είναι η σύμβαση αυτή της Κωνσταντινούπολης και παρόλα αυτά, παρόλο που είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μα για να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και την ενδοικογενειακή βία, γιατί και περί αυτής πρόκειται, παρόλα αυτά δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά οι κυβερνήσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της δεν έχουν φροντίσει να βιαστούν για να γίνει αυτή η επικύρωση της σύμβασης τους Κωνσταντινούπολη. Οπότε με μικτά συναισθήματα, ικανοποίηση από τη μία και απογοήτευση από την άλλη, έχω εμπιστοσύνη στο έργο μας και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε έγκαιρα η προηγούμενη Προεδρία δεν τα κατάφερε. Αυτή η Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοντεύει να τελειώσει τη θητεία της και δεν είμαι και σίγουρα αν θα τα καταφέρει. Πρέπει τέλος πάντων να κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η σύμβαση αυτή της Κωνσταντινούπολης και όλοι μετά θα μπορούμε με ένα τόσο σημαντικό εργαλείο, τόσο ισχυρό, να απαλείψουμε αυτό το φαινόμενο που μας ντροπιάζει όλους ως δημοκράτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπλιμπάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και τη Κριστίν και την Άννα Μαρία για τη δουλειά τους και για τη συμμετοχή τους ε, στην Επιτροπή. Εγώ νομίζω ότι στην πολιτική ένα μέρος ε, της δουλειάς μας μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανος και αυτό είναι ένα από τα ιστορικά βήματα και σίγουρα θα είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή μας ε, Φαίνεται εντυπωσιακό πως ε, όταν ε, υπάρχουν θύματα και τα θύματα είναι γυναίκες, ε, να μην υπάρχει πολιτική αντίδραση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως όλοι μας τα περιμέναμε να συμβαίνει καθημερινά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Εδώ και τρία χρόνια έγινε η πρώτη έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα δείγμα με διάφορες συνεντεύξεις που ελήφθησαν από Ευρωπαίες γυναίκες. Δεν θα τα επαναλάβω τα αποτελέσματα, γιατί είναι πραγματικά ανησυχητικά, δραματικά. Σήμερα έχουμε ε, το χάρη μια επίθεση και ε, τελικά μπορεί να έχουμε νεκρούς ε, και όλοι ε, φυσικά αντιδρούμε, γιατί είναι κάτι απαράδεκτο, όμω δεν αντιδρούμε καθόλου στη βία κατά των γυναικών και έχουμε καθημερινά θύματα γυναίκες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πει απαιτούμε, υποχρεώνουμε το Συμβούλιο να κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να γίνει. Θα αρκούσε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ακόμη, εγώ δεν είδα ούτε ένα καν επιχείρημα γιατί τα κράτη ε, δεν θέλουν να κυρώσουν και γιατί δεν δέχονται αυτή τη σύμβαση, γιατί δεν δέχονται το περιεχόμενο τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ασκούν την επαρκή πίεση σε όσους δεν θέλουν να κυρώσουν για να τους πούν είναι απαραίτητο. Πώς θα μιλήσουμε για τις ευρωπαϊκές αξίες αν δεν είμαστε ικανοί να γνωρίσουμε αυτή τη βία. Λεχθέντως αυτού, νομίζω ότι πράγματι θα έπρεπε να αναφέρουμε αυτό να γίνεται αναφορά και στη βία κατά των γυναικών με αναπηρία, γιατί ε, φυσικά είναι η ομάδα που υποφέρει περισσότερο από τη βία και να γίνει και μια ειδική μνήμα στα παιδιά. Όταν μιλάμε στα γόρια και στα κορίτσια για γυναίκες που υφίστανται έμφυλη βία, μας λένε δεν δίνεται παρκής προσοχή στα κορίτσια και στα γόρια γυναικών που υποφέρουν από οικογενειακή βία, γιατί φαίνεται να είναι το τμήμα της βίας που είναι το πιο κρυφό. Νομίζω λοιπόν ε, ότι θα πρέπει να κάνουμε μια εξωτερική και χρειαζόμαστε και στατιστικά στοιχεία γιατί υπάρχουν χώρε όπου θεωρούν ακόμη ότι η βία κατά των γυναικών είναι μέρο τη ιδιωτική ζωή και δεν είναι δημόσιου χαρακτήρα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν περισσότερε εκστρατείε, περισσότερη ευαισθητοποίηση. Και τέλο. Θα πρέπει να αναφέρουμε την ανάγκη να εργαστούμε στο πεδίο της πρόληψης. Για να προλάβουμε θα πρέπει να έχουμε μια πολιτιστική αλλαγή, θα πρέπει να προχωρήσει η πολιτική συνδυτοποίηση χρειάζεται εμπλοκή σε τοπικό επίπεδο, γιατί η εμπλοκή σε τοπικό επίπεδο και οι συμφωνίες μας επιτρέπουν να προχωρούμε και έχουμε βέλτιστες πρακτικές που μας το δείχνουν αυτό. Και θα κλείσω λέγοντας, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να πιέσουμε προς τα πάνω για να ακυρωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά νομίζω ότι χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες επειδή δεν έχουμε ένα θεματολόγιο, ένα τόπο που να καταγράφονται όλες οι καλές πρακτικές ευρωπαϊκό επίπεδο για να χρησιμεύουν ω παράδειγμα για τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να στραφώ στις δύο συγκίτρες. Να ξεκινήσω με την Κριστίν. Ευχαριστώ πολύ. Όλου όσου πήραν το λόγο. Πραγματικά οι παρεμβάσει σα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μπιλμπάο, τον περασμένο Νοέμβριο όταν ψηφίσαμε, όταν ευθετήσαμε αυτό το ψήφισμα, πρόκειται για ένα κοινό ψήφισμα πρακτικά όλων των ομάδων του Κοινοβουλίου. Ακριβώς αυτό κάναμε. Θέλουμε να ζητήσουμε τα κράτη να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη σύμβαση και επίσης τους ζητήσαμε να προχωρήσουν σε αυτή την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ε, χρειάζεται χρόνος. Ακούσαμε ότι κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ε, ότι αυτό θα φερούσε μεγάλο μέρος τη κυριαρχία τους. Ε, εγώ θέλω να πω ότι η βία κατά των γυναικών δεν έχει σύνορα. Πρέπει να μπορούμε να προστατεύουμε τις γυναίκες όπου και να βρίσκονται εντός της Ένωσης. Και τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να φοβούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει, δεν ε, είναι κατά των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Άκουσα και όσο είπε η κυρία Στίβενς ε, και ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να θεωρηθούν ευάλωτα. Ναι, το διευκρινίζουμε αυτό ε, στην έκθεση, το ίδιο και για τους ΛΟΑΔ. Εδώ θέλω να σας πω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, εντελώς απαράδεκτες πρακτικές. Σε ό,τι αφορά τώρα την Πολωνία και το γεγονός ε, ότι θα μπορούσε κάποιο κράτος ε, μέλος όταν έχει κυρώσει τη σύμβαση δεν μπορεί να επανέλθει, να χωρίσει, ναι βεβαίως. Εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε την υπογραφή, την κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ρήτρα γέφυρα είναι ένα σημαντικό στοιχείο που ενεργοποιείται εδώ. Έχουμε λοιπόν το θέμα του χρόνου. Η ανταλλαγή βαλτίστων πρακτικών είναι κάτι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκες και κορίτσια που πεθαίνουν. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα νομικό εργαλείο, υπογραφή της σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρό νομικό εργαλείο και η οδηγία θα είναι ακόμη περισσότερο. Η ανταλλαγή βαλτίζων πρακτικών και συζητήσει ε, δεν εμπαδίζουν ε, το θάνατο των γυναικών μέρα με τη μέρα. Ευχαριστώ, Ιάννα Μαρία. Ευχαριστώ πολύ και ε, είμαι ευγνώμων για όλη την υποστήριξη από την πλευρά των συναδέλφων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό που το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε φωνή στις εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών που υποφέρουν ε, σιωπήρα και να τους δείξουμε ότι δεν είναι εγκαταλειμμένες ε, και να δείξουμε την αποφασιστικότητα ανεξαρτήτως των πολιτικών μας κομμάτων και απαιτείται συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Όπως είπε η κράτη-μέλη, χρειάζεται διάλογο, δείχνοντας σεβασμό προ τι διαφορετικές διαφορές, ε, τις ανησυχίες, ε, τις ε, καταστάσεις που μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε κράτο μέλο, κράτος μέλος, χωρίς όμως αυτό να δικαιολογεί ότι δεν θα κάνουμε τίποτα για να καταπολεμήσουμε τη βία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαλτέζικη Προεδρία διότι έχουμε λάβει μεγάλη υποστήριξη ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο που ήμασταν εκεί για την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ε, και είχαμε μία συνάντηση μεταξύ της Προεδρίας, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και αυτό ίσως να είναι συμβουλικό, όμως ταυτόχρονο δείχνει ότι οι τρεις θεσμοί συνεργάζονται το, ε, η επιθυμία ε, κάποιων ε, κρατών μελών να ε, υπαναχωρήσουν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επικοδομητικό τρόπο. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω κάποια σχόλια από συναδέλφους. Ναι, αρκετά ζητήματα δεν έχουν συμπεριληφθεί λόγω χώρου, ότι θα το κάνουμε αυτό με τις τροπολογίες ε, και ε, κυρία Στίβενς ε, κάνουμε, διοργανώσαμε μαζί μια συνάντηση και συζητήσαμε, προεδρεύσαμε μαζί σε μια συζήτηση για τα παιδιά με αναπηρία και σίγουρα θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε αυτό διότι ε, η ε, παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι παραβίαση θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και θα πρέπει να αυξήσουμε την ενημέρωση για αυτό. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και αυτό είναι το πιο σημαντικό ε, για την ε, σύμβαση. Δεν αφορά μονάχα την τιμωρία, αλλά την ε, μακροπρόθεσμη εργασία για την ενίσχυση των γυναικών. Ναι, η πλήρη εφαρμογή αναφέρεται στο κείμενό μας και αυτό θα το τονίσουμε ιδιαίτερος, διότι είναι το πρακτικό κομμάτι. Και Μαρία Γκαμπριέλα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την υποστήριξή σου. Γνωρίζω τις δυσκολίες και θα ήθελα να σου πω ότι εμείς στο ΕΛΚ έχουμε μια ε, ε, πρακτική προσέγγιση στην μηδενική ανοχή. θα πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένους ε, τρόπους ε, για να αναφερθούμε στις ανησυχίες των μελών. Σε μια κρόαση πριν από μερικές εβδομάδες της Επιτροπής ΦΕΜ προσκαλέσαμε μια σου ειδική οργάνωση και ε, συγκεκριμένα όσον αφορά αυτό που αναφέρατε εσείς ε, Άννα Μαρία ε, παρουσίασαν το πώς μπορεί να γίνει η εργασία με ψυχολογική υποστήριξη, με κατευθυντήριες για να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη και να μπορέσουν να παράσχουν εκπαίδευση, ε, περίθαλψη. Έτσι λοιπόν μπορούμε από αυτή τη συζήτηση να πάμε σε συγκεκριμένη δράση για να δείξουμε στα κράτη-μέλη το τι μπορούν να κάνουν και ναι, ε, παντού, ακόμα και ε, αγόρια ε, στον ιδιωτικό τομέα. Είπαμε ότι θα πρέπει να, να αναφερθούμε σε νέα είδη βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, την εκδικητική πορτογραφία, αλλά και άλλες μορφές εγκλημάτων, για τα οποία δεν είχαμε το χώρο να τα τοποθετήσουμε στο κείμενο, όμως θα το κάνουμε μέσω των τροπολογιών. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι υποστηρίζω την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγνωρίζω ότι το ποινικό δίκαιο είναι ένα εθνικό ζήτημα, όμως χρειαζόμαστε κοινά δεδομένα, χρειαζόμαστε ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε ε, τις ικανότητες των κρατών για να αντιμετωπίσουν αυτή τη βία το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας ε, και αδειμονώ στην μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ την κυρία Κοράσα Μπίλτ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το χρονοδιογράμμα για την κατάθεση ε, τροπολογιών είναι η 26 Απριλίου στις 5 το απόγευμα. Να λάβετε υπόψη σας όμως ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν θα είναι σε μορφή 84am ε, διότι έχουμε να κάνουμε ε, για μια ε, νομοθετική διαδικασία συνένεσης. Θα τα καταθέσετε αυτά στη θηρίδα ενώ η γραμματεία θα σας αποστείλει ένα mail με αναλυτικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα στην κοινή Σας Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, και ε, την Πρόεδρο αλλά και τα αξιότιμα μέλη της ΦΕΜ και θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη ε, της ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Um, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα καθώς οι συνάδελφοι της ΦΕΜ αποχωρούν.